Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στην τελική μας φάση και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία μέχρι το τέλος του έτους. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν. Φαντάζομαι ότι έχετε μία επιπρόσθετη ερώτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ το Συμβούλιο για την απάντησή του. Ιδιαίτερα χαίρομαι που λέτε ότι θα μπορούσε να διεκπαιρωθεί το θέμα από το τέλο του έτου, διότι νομίζω ότι είχατε πει ότι 16, 13 είπατε εσεί. εγώ έλεγα 16 κάτι μέλη έχουν κυρώσει το Συμβούλιο. Μπορεί να μου πει ποιες ήταν οι συνέπειες όσον αφορά την ε, επικύρωση πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως αυτής της συμβάσεως. Αναφέρατε κάποια άρθρα. Προφανώς υπάρχουν κάποια άρθρα που εμπεριέχονται στη συμβασή. Άρθρα που αναφέρονται στο θέμα της λογικής ε, ε στέγασης ανθρώπων με ειδικέ ανάγκε το δικαίωμα να ζουν ανεξάρτητα. Ποια συνέπεια θα είναι αυτού. Το ερώτημά μου είναι, ποια θα είναι αντίκτυπο τη του πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώσεω αυτή τη σύμβαση επί των χωρών εκείνων που δεν την έχουν επικυρώσει. Σα ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, επανέρχομαι επί ενό στοιχείου. Πρόκειται περί 13 κρατών μελών που επεκύρωσαν την σύμβαση. Θέλετε να σας παραθέσω τις χώρες για να μαστιγώσει ότι τους δε, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία επεκύρωσαν αυτή την σύμβαση. Ποια είναι η κατάσταση τώρα. Βεβαίως πρέπει να αναμένεται μια συμφωνία σε αυτό κώδικα ε, ε, ε, για μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν κατατεθεί το μέσο επίσημης επικύρωσης που θα ολοκληρώσει την κύρωση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως της Συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών που αφορά τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν κάποια αναπηρία. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Λοιπόν, η επικύρωση τη συμβάσεω θα ολοκληρωθεί και μετά το Συμβούλιο θα μπορεί να επανέλθει στο θέμα ενδεχόμενη εργαλειοθήκη για ενεργό προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Μια ιδέα που προτάθηκε εξάλλου από πολλά κράτη-μέλη. Ε, και έγινε δουλειά προ αυτό το θέμα παράλληλα με την προετοιμασία πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στατική για την Ευρωπαϊκή Ένωση 2010-2020 για τα άτομα με αναπηρία. Αυτή η στρατηγική θα προβλέπει σχέδιο δράσης για την επόμενη δεκαετία με στόχο την εγγύηση τα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν πλήρως των δικαιωμάτων τους και των ελευθεριών τους. Σας ευχαριστώ. Έχω και άλλε δύο συμπληρωματικέ ερωτήσει. Η μία θα ακολουθήσει την άλλη. Και μετά, κύριε Υπουργέ, θα σα παρακαλέσω να απαντήσετε και στι δύο. Ο κύριο Ζέμκα και η κυρία Μπρίνκεβιτσιούτε. Ευχαριστώ. Κυρία Ντέγκα πρώτα. Ο κύριος Ντέγκα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν επιτρέπετε θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα κυρία Υπουργέ. Ένα ερώτημα σημαντικό κατά την άποψή μου. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ κακή διότι από τα 27 κρατημέλη μελη 13 μόνο έχουν κυρώσει αυτή τη σύμβαση. Τα περισσότερα κράτη, τα 14, δεν έκαναν κάτι τέτοιο ακόμα. Ερώτημα το εξή. Γνωρίζετε τους λόγους για τους οποίους μόνο τα μισά κράτη-μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση που είναι πάρα πολύ σημαντική για τα άτομα με αναπηρία. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Μπλινκεβιξιούτε έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για την ε, απάντησή σας. Θα ήθελα να γνωρίζω για ποιο λόγο τα κράτη-μέλη δεν βιάζονται τόσο να επικυρώσουν αυτή τη σύμβαση του ΟΗΕ. Φοβούνται να επομιστούν τις ευθύνες τους. Όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία. Η οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων ε, λήφθη υπόψη παρκώς. Πώς πάνε οι δουλειές, πώς, πάει, πώς πάνε οι προσπάθειες. Μπορεί, μπορεί τελικά αυτή η οδηγία να επιταχυνθεί και να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με τα κρατη να προχωρήσει τα πράγματα πιο γρήγορα. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ακούστε. Οι εργασίες ε, ουσιαστικά γίνονται ε, σε επίπεδο κρατών μελών αν μου επιτρέπετε μπορώ να πω ότι πράγματι μπορεί κανείς να εκφράσει την απογοήτευσή του ή το σκεπτικισμό του ό,τι αφορά ε, την καθυστέρηση ακριβώς επικύρωσης ε, για κάποια κράτη-μέλη. 13 επαναλαμβάνω αυτά τα οποία έχουν ε, προβεί στην επικύρωση. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Νομίζω ότι απλά ο τρόπο με τον οποίο επικυρώνουν τα κράτη-μέλη ε, ακολουθεί διαδικασίε που μπορεί να διαφέρουν από το ένα κράτο μέλο στο άλλο. Δεν θέλω να επεκφύγω ούτε να κρυφώ πίσω από το επιχείρημα αυτό, αλλά πρέπει να πω επίση ότι και σε αυτό το τομέα, όπω και σε άλλου υπάρχει κάποια εθνική κυριαρχία στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο προχωρούν τα κράτη-μέλη στην επικύρωση. Φυσικά μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να κινηθούν γρηγορότερα, θα μπορούσαν ήδη από την αρχή να συνεργάζονται περισσότερο μεταξύ τους τα κράτη-μέλη, πάντως για ορισμένα ζητήματα τίθεται το θέμα αυτό ακριβώς της εθνικής κυριαρχίας. Η πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Την είχε καταθέσει αρχικός ο κύριος Μίτσελ. Σήμερα όμως θα εκπροσωπηθεί ο κύριος Μίτσελ από την κυρία Μακγκίνες. Ε, αφορά η ερώτηση τη θεραπεία της επιληψίας. Έχετε το λόγο όταν είστε έτοιμος κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, αν και απόντα, τον ε, κύριο βουλευτή που κατέθεσε την ερώτηση αυτή και για το ενδιαφέρον του βέβαια για το ζήτημα αυτό σίγουρα οι νευροεκφυλιστικές νόσοι, οι εγκεφαλικές, ε, μη ψυχιατρικές νόσοι, των οποίων δηλαδή και η επιληψία, είναι μείζον λόγος ανησυχίας και πλήττουν αρκετούς ε, πολίτες μας. Με βάση το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της δημόσιας υγείας και της πρόληψης ασθενειών. Επομένως, η προσέγγιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οριζόντια και επικεντρώνεται στην καταπολέμηση του στίγματος και της αρνητικής διάκρισης κατά ατόμων με νευροεκφυλιστικές νόσους, ε, εγκεφαλικά νοσήματα μη ψυχιατρικού τύπου και γι' αυτό στα συμπεράσματά του το Συμβούλιο σε αφορά την καταπολέμηση της διάκρισης ε, και του ε, στίγματος είχε ζητήσει από τα κράτη-μέλη να δώσουν προσοχή συγκεκριμένα σε αυτά τα ζητήματα που οδηγούν στο στιγματισμό αυτών των ατόμων και πρόκειται άλλωστε για κάτι που αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες. Πρέπει να αναγνωριστεί αυτό το πρόβλημα και να του δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη μείωση του κινδύνου αποκλεισμού, κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων αυτών. Στις 3 Ιουνίου 2005, στα συμπεράσματα σχετικά με μια κοινοτική δράση για τον τομέα της ψυχικής υγείας, ε, το Συμβουλίο κάλεσε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν στην πράξη αυτή τη διακήρυξη καθώς και το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Υπουργικής Διάσκεψης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την ψυχική υγεία. Ε, η συνάντηση αυτή είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2005 στο Ελσίνκι. Τέλος, το Συμβούλιο έχει δεσμευθεί ιδιαίτερα ε, στον αγώνα κατά μιας άλλης εκφυλιστικής νόσου, προβλημάτων νευρολογικών, ε, νευρολογικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα πρόκειται για την νόσο του Αλτσχάιμερ. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2008 ε, μιλήσαμε για τη στρατηγική καταπολέμησης νευροεκφυλιστικών νόσων σχετιζόμενων με την γύρανση και δι για την νόσο του Αλτσχάιμερ. Και στη, στα συμπεράσματα τη 3η Δεκεμβρίου 2009 για την κοινή προετοιμασία, για την κοινή έρευνα στην Ευρώπη ε, που καλύπτει ιδιαίτερα πιλωτικές ε, δράσεις για την καταπολέμηση νευροεκφυλιστικών νοσημάτων και δι την νόσο του Αλσχάιμερ. Thank you very much, Mrs. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, Συμβούλιο, για την απάντησή σας και θα διαβιβάσω την εκτίμηση αυτή που εκφράσατε στη συνάδελφο. Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών. Κάτι που πρέπει να απασχολεί το Συμβούλιο. Για την επιληψία υπάρχει διαφορά ανάλογα από το που μένει κανεί. Και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα την έλλειψη νευρολόγων σε κάποια κράτη-μέλη. Θα μπορούσατε επίση να ασχοληθείτε και με το θέμα τι συνέπειε έχει αυτό για τη συνοριακή περίθαλψη και το σχετικό πακέτο το οποίο συζητείτε διότι αν δεν θεραπεύεται υποφέρουν σε μεγαλύτερο ποσοστό οι άνθρωποι από ότι αν υπάρχει επαρκής θεραπεία. Και είναι λυπηρό το ότι υπάρχει διαφορετικό επίπεδο φροντίδας στις διάφορες χώρες μέλη για τους ανθρώπους που πάσχουν από επιλήψη. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ το λόγο για να απαντήσετε. Λοιπόν, νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο στη διαπίστωση που εκφράσατε δηλαδή την ποιοτική πτυχή την ιατρική που αφορά τα διάφορα κράτη-μέλη. Ποιοτικά έχουμε πόρο από εναρμόνιση της περίθαλψης, της υγείας, του τομέα της υγείας. Όσον αφορά την υγεία, τα εξουσίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι πολύ μικρές σε σχέση με την εθνική αρμοδιότητα και καλά κάνετε που αναφέρεστε στο διασυνοριακό αυτό πακέτο διότι προφανώς πρόκειται περί στοιχείου το οποίο δύναται να βελτιώσει κάποιες ποιοτικέ πτυχές όσον αφορά την περίθαλψη. Επί Βελικής Προεδρίας υπενθυμίζω ότι το Συμβούλιο συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις, θα συνεχίσει μέχρι τέρμα με στόχο να ε, συντονιστούν οι απόψεις για να καταλήξουν δεύτερη ανάγνωση συμφωνία όσον αφορά το πακέτο αυτό που συνδέεται με την διασυνοριακή περίθαλψη. Δύσκολο εγχείρημα, περιορισμένος ο χρόνος αλλά έχουμε τη φιλοδοξία να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα πριν το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Δεν έχω επιπρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα αυτό και προχωράμε στην επόμενη η οποία προέρχεται από τον κύριο Κέλλη και αναφέρεται στο συντονισμό της θέσης της Ευρωπαϊκής Ενώσης στο Κανκούν. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Συμβούλιο στην συνεδρίασή του της 14ης Οκτωβρίου υιοθέτησε συμπεράσματα για την θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την διάσκεψη στο Κανκούν για το κλίμα όπου θα πρέπει να εξετάσουμε το γενικό πλαίσιο όσον αφορά τις κλιματολογικές αλλαγές όπου στο Συμβούλιο ε, του Οκτωβρίου που θα γίνει 18 και 19 Οκτωβρίου θα θα οριστεί η θέση 28 και 29 με Οκτωβρίου θα διευκρινιστεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η οποία αναφέρεται σε όλα τα βασικά θέματα σχετικά με αυτό το συνέδριο τα προσδοκόμενα αποτελέσματα την επέκταση της ε, συμφωνίας του Κιώτο πέραν του 2012 τα ε, θέματα τα οποία περιλαμβάνει το χάρτης πορείας του Μπαλί η προστασία των δασών, των τεχνολογιών και τη χρηματοδότηση. Γι' αυτό και το Συμβούλιο προσπάθησε να διατυπώσει σαφείς θέσεις οι οποίες να μπορούν να, επι, ε, ε, ε, να μεταφερθούν εύκολα. Και τώρα θα πρέπει να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα και στους διεθνείς ομολόγους μας όπως το ανέφερε το Συμβούλιο διότι ελπίζουμε ότι στη συνεδρίαση του θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε μία ισορροπημένη, ένα ισορροπημένο σύνολο αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο για να προστατευτεί το κλίμα μετά το 2012. Πολλές ε, συναντήσεις και διμερείς επαφές θα γίνουν πριν από το Κανκούν και θα δώσουν τη δυνατότητα να εξηγήσουμε στους συναδέλφους τη θέση μας και στη διάσκεψη οι θέσεις αυτές θα διευκρινιστούν στις συνεδριάσεις συντονισμού που θα οργανώνει τακτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως ελπίζουμε ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα συμβάλλουν στο στόχο αυτό μεταδίδοντας αυτό το μήνυμα σε όλες τις εξωτερικές επαφές τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι τη θέση σας και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όντως να έχουμε μία θετική επίπτωση στο Κανκούν ε, και όχι όπως ατυχώς έγινε στην Κοπενχάγη. Θα ήθελα να κάνω μία επιπρόσθετη ερώτηση. Αντιλαμβάνομαι ότι ε, ε, ε, εφόσον ε, έχετε το παράδειγμα της Κοπενχάγης πόσο δεσμευτική πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η έκβαση της διασκέψεως στο Κανκούν για τη μελλοντική κατάσταση. Λοιπόν, πρέπει να σας πω και να διευκρινίσω ότι όντως η πρόοδος θα είναι δύσκολη στο Κανκούν για τρεις λόγους γιατί είμαι σχετικά απεσιόδοξος καταρχήν λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πολλές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και όπου καταλήγουμε ότι οι καλές προθέσεις ε, για επενδύσεις ε, ε, επί του θέματος είναι μάλλον πιο περιορισμένες. Επίσης όλο και λιγότεροι θέλουν να αναλάβουν δεσμευτικές υποχρεώσεις και απέτυχε στις Ηνωμένε Πολιτείε η οθέτηση μια σαφής, σαφούς νομοθεσίας επί του θέματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διατηρήσει στις τις θέσεις που διατύπωσε στην Κοπενχάγη και πρέπει να προσέχουμε με ποιο τρόπο τώρα δεσμευόμαστε για να μην υπονομεύσουμε τις θέσεις τις οποίες θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουν στο Κακούν σε ένα μήνα. Ευχαριστώ. Ε, η πρόσθετη ερώτηση από αυτού έχουν ζητήσει διάφοροι αλλά θα δεχτώ δύο για να υπάρχει πολιτική ισορροπία πρώτα από την κυρία Τικάου και μετά του κυρίου Όμπερμάιερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Προτίθεστε να σχετίσετε τους στόχους για την κλιματική αλλαγή μείωση της ρήπανσης δηλαδή, με τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Αληθεύει πράγματι ότι υπάρχουν αναπτυσσόμενες χώρες που πιστεύουν ότι είναι πάρα πολύ δαπανηρό για αυτές να περάσουν σε ένα ποσοστό περιστολής των εκπομπών και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ε, νέες ε, περικοπές ή μείωση και δεν ξέρουμε αν θα βοηθήσει την βιώσιμη οικονομία. Λοιπόν, θα συσχετίσετε αυτό με τους αναψυκτικούς χιλιετίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην Κοπενχάγη ακόμη και συνεργαζόμενες χώρες όπως η Ινδονησία και η Βραζιλία ε, συμφώνησαν σε ένα μπλοκ έναντι των χωρών του Βορρά και πρόκειτο για, ένα, ε, για μια συζήτηση δικαιοσύνης και φαντάζομαι ότι στο Κανκούν δεν πρόκειται να προβούν σε υποχωρήσεις οπότε πώς μπορούμε υπό αυτά κατάσταση συνθήκας να ε, φύγουμε μία αποτυχία και τι θα γίνει με τα θέματα αυτά εάν δεν αναλάβει ένα μεσολαβητικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, για να απαντήσω στα δύο ερωτήματα αυτά, πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι έχετε δίκιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει στρατηγική εναντί τη Κοπενχάγη. Θα πρέπει να εξηγήσει πολύ καλύτερα τη θέση τη θα πρέπει να συνομιλήσει με ομάδες χωρών που έχουν ε, αρκετά διαφορετικές απόψεις από τις δικές μας και πράγματι η διασύνδεση αλλαγής του κλίματος και στόχου της χιλιετίας και στόχων της χιλιετίας έχουν, υπάρχει διασύνδεση προφανής. Δεν μπορούμε να ζητάμε τα επόμενα χρόνια την ίδια προσπάθεια από εκείνους που πρέπει να μειώσουν μεγάλο παθητικό βιομηχανικό όπως εντός της ενώσεως και από τις χώρες που αναπτύσσονται. Εξάλλου γι' αυτό φαίνεται να μην φτάνει, αλλά γι' αυτό όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει σημαντικά στην αρχή, στην, αρχή του Fast Arc, ενίσχυση των χωρών των αναπτυσσομένων και αυτό το μέτρο στοχεύει στις χώρες που δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα για να πετύχουν τις δέωσες μειώσεις. Αποτελεί ένα σύνολο. Ο διάλογος και τα προσαρμοσμένα μέσα θα πρέπει να μπορέσουν τελικά να επιτρέψουν έναν ενδελεχέστερο προβληματισμό από πλευρά αναπτυσσομένων χωρών όσον αφορά του ίδιου του στόχου που έχουν για την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Σας ευχαριστώ. Θα πάμε στο επόμενο ερώτημα του κυρίου Παπα-Νικολάου και αφορά το πρόγραμμα της Προεδρίας και την, ε, όταν, την πρόορη αποχώρηση από το σχολείο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, η Προεδρία ακολουθώντας τις εργασίες που ξεκίνησε η πρώτερη Προεδρία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Συνεργασία, όσον αφορά την σχολική ε, εκπαίδευση, δίνει ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τις βασικές αρμοδιότητες και όσον αφορά την εγκατάλειψη του σχολείου και δίνει συνέχεια στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2010 που υπογράμμισε εκεί την ανάγκη της μείωσης του ποσοστού της, σχολικής, της πρόορης σχολικής εγκατάλειψης στην Ευρώπη και να καθορίσει ένα γενικό στόχο αυτό το ποσοστό να κατέβει κάτω από το 10% μέχρι το 2020. Στα πλαίσια αυτής της προοπτικής η Προεδρία ξεκίνησε διάφορες πρωτοβουλίες, ξεκινώντας από το σεμινάριο υπουργικού επίπεδου που διοργάνωσε αρχές της θητείας της τον περασμένο Ιούλιο αυτό το σεμινάριο καθώς και συνεδρίαση των Γενικών Διευθυντών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που προηγήθηκε την παραμονή εξέτασαν την δυσκολία απόκτησης βασικών ε, προσόντων ε, μαθηματικά, επιστήμες, μετρική γλώσσα και την εμπειρία που έχουν τα κράτη-μέλη και ποιοι είναι οι πολιτικοί προσανατολισμοί που θα πρέπει να ακολουθηθούν και να αναπτυχθούν όσον αφορά την πρόληψη αυτής της πρόληψη σχολική εγκατάλειψης. Μετά από αυτή τη συνεδρίαση η Προεδρία επεξεργάστηκε συμπεράσματα σχετικά με τη σημασία που έχει να αυξηθούν οι βασικές δεξιότητες στα πλαίσια της ευρωπαϊκής συνεργασίας, στα πλαίσια της σχολικής εκπαιδεύσεως. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο όσον αφορά αυτά τα συμπεράσματα έχουν δρομολογηθεί θα μπουν στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου του επομένου Νοεμβρίου. Αυτό προβλέπει η Προεδρία. Γενικότερα τώρα το Συμβούλιο τελεί ένα αναμονή προτάσεως συστάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα πρέπει να υποβληθεί προσεχώς όσον αφορά το πρόβλημα αυτό τη ε, πρόορη σχολική εγκατάλειψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν και σε εθνικό επίπεδο οι προσπάθειε, ούτω ώστε να μειωθεί σταδιακά το ποσοστό αυτό τη πρόορη σχολική εγκατάλειψη μέχρι το 2020 σύμφωνα με τους στόχους που καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για να κλείσω, θα επισημάνω επίσης ότι το πλαίσιο τη Ευρωπαϊκού έτους για την καταπολέμηση τη φτώχειας και του νοικού αποκλεισμού. Σε αυτό το πλαίσιο η Βελική Προεδρία διοργάνωσε στις 28 Σεπτεμβρίου που μας πέρασε τη διάσκεψη με τίτλο «Να σπάσει ο φαύλο κύκλο της ανισότητας και πώ θα επιτεθεί κοινωνική ένταξη μέσω τη εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα αυτή τη διασκέψη θα τροφοδοτήσουν την ανταλλαγή απόψεων που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Παιδεία που θα λάβει χώρα την 19η Νοεμβρίου. Σα ευχαριστώ, ρε, Πρόεδρο. Ο κ. Παπα-Νικολάου, έχετε κάποια συμπληρωματική ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την απάντησή σα. Στα όσα μα είπατε, θέλω να προσθέσω τα εξή ερωτήματα. Όλα αυτά τα παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο πού πάνε μετά στο περιθώριο στον κοινωνικό αποκλεισμό ή σε κάποιο τεχνικό επάγγελμα που αυτό είναι μια καλή εξέλιξη που τους εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή διαβίωση. έχει στη διάθεσή του το συμβούλιο κάποια σχετικά στοιχεία ή τουλάχιστον έχει ζητήσει ή σχεδιάζει να ζητήσει από την επιτροπή να κάνει αυτό που ονομάζουμε χαρτογράφηση των κοινωνικών διαδρομών προκειμένου να ξέρουμε ποια είναι η συνέχεια της ζωής αυτών των παιδιών και πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις πολιτικές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ συνάδελφε, η πρωτοβουλία είναι εξαιρετική και πρέπει να σας πω επίσης ότι οι επαφές μεταξύ υπουργών ε, ε, και ανωτάτέρων αξιωματούχων ε, των Υπουργείων Παιδείων μας δείχνουν ότι η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από τη μια χώρα με στην άλλη. Υπάρχουν προγράμματα ορισμένες προς τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα σε ορισμένες χώρες ώστε αυτοί οι οποίοι εγκαταλείπουν το σχολείο να μην περιθωριοποιηθούν αυτή η χαρτογράφηση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βέβαια, θα απαιτηθεί χρόνος, γιατί η αξιολόγηση της κατάστασης στα 27 κράτη-μέλη, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Νομίζω ότι ξεκινούμε τις εργασίες για την ε, πρόορη σχολική εγκατάλειψη επί Βελγικής Προεδρίας. Θα συνεχιστούν ε, όμως οι προσπάθειες αυτές επί Ουγγρικής Προεδρίας που φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει και ένα σχέδιο σύστασης όχι μόνο για την μείωση του ποσοστού της πρόορη σχολικής εγκατάλειψης αλλά και για να καταλήξει και σε ό,τι αφορά αυτή τη χαρτογράφηση ε, στις 27 χώρες μέλη για να δούμε τι απογίνεται με αυτούς τους ε, μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο και ιδίως όταν αυτοί περιθωριοποιούνται και δεν στρέφονται, όπως είπατε, στην τεχνική εκπαίδευση, για παράδειγμα. Thank you. Again, I have... Uh, Ευχαριστώ και πάλι έχω δύο συμπληρωματικά ερωτήματα. Μπλινκεβιτσιούτε και Τικάου. Η κυρία Μπλινκεβιτσιούτε. Πρώτα αυτή τη φορά. Εκτός μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ. Οι προσπάθειες της Βελγικής ε, Προεδρίας σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ε, φτώχειας είναι σημαντικές. Σε πλαίσιο της προσπάθειας αυτής δεν θέλω να σα ρωτήσω, δεν θεωρείτε ότι συμβάλλει η φτώχεια ακριβώς και στην προορισχολική σχολική εγκατάλειψη. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτησε ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα mm. για το κατώτατο εισόδημα στις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν πιστεύετε ότι η καταπολέμηση της φτώχειας θα μπορούσε, θα μπορούσε με αυτό το μέτρο διακόπτει δυστυχώ η πρόεδρος, η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Δυστυχώ το ποσοστό της σχολικής εγκατάλειψης ανέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 19% και σε χώρες ε, που υπάρχει πρόβλημα με τη φτώχεια οδηγεί και στο κλείσιμο σχολείων, ιδίως στην Ήπεθρο. Όταν μιλάμε για την παιδεία, για την εκπαίδευση, μιλάμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φέτος που έχουμε το έτος καταπολέμησης τη τόκης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σα παρακαλέσω να θέσετε υποχρεωτικού στόχου για τη μείωση τη σχολική εγκατάλειψη. Πρώτα σας ευχαριστώ και τους δύο, και τις δύο μάλλον, ο Υπουργός έχει το λόγο. Συμφωνώ και με τις δύο παρεμβάσεις γιατί όντως όποιος εγκαταλείπει το σχολείο οδηγείται στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι προφανές ότι πολλά παιδιά λόγω οικογενειακής προελεύσεως, οικονομικής προελεύσεως και καταστάσεως των γονέων δεν βοηθούνται ε, από την οικονομική κατάσταση και ε, το φαινόμενο αυτό διονγκώνεται. Το αντελήφθη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι όπως ξέρετε από κοινού υιοθετήσαμε τη στρατηγική για το 2020 η οποία ε, συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη, την ποιότητα της εκπαιδεύσεώς μας και την καταπολέμηση της φτώχειας για να αποτελέσουν ένα σύνολο που επιτρέπει να απαντήσουμε συνεκτικά στο πρόβλημα δεν θα επανέλθω στις αρμοδιότητες κλειδιά παρόλο που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα υποβάλει η Βελγική Προεδρία στο Συμβούλιο του Νοεμβρίου. Θα τα αναφέρω όμως εντάχει. Εθνική στρατηγική για να βελτιωθεί η απόδοση των μαθητών εις το διάβασμα στην ανάγνωση αλλά και στις ανταλλαγές. Μία εθνική στρατηγική για να υπάρχει υπάρχει μία τράπεζα δεδομένων κατά τρόπον ώστε να μπορεί κανείς ε, να λάβει τις σωστές αποφάσεις και συνειδητοποίηση στα κράτη που το επιθυμούν της καταστάσεις για να βελτιωθούν οι βασικές γνώσεις των νέων Ευρωπαίων και καλύτερη χρησιμοποίηση των ε, μέσων που διαθέτουμε σαν την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, το πρόγραμμα της εκπαιδεύσεως, διαβίου μάθηση και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την τεχνολογική ανάπτυξη. Ορισμένοι ε, από τους ε, ε, στόχους που έχουμε είναι αυτοί και η Βελγική Προεδρία και οι επόμενες, συγκεκριμένα μάλιστα η Ουγγρική Προεδρία, θα συνεχίσουν αυτό το έργο. Ευχαριστώ. Τώρα προχωράμε στην ερώτηση του κυρίου Χίγκινγκ που αναφέρεται στο στόχο της Ευρωπαϊκής Ενάωσης για την πλήρη εξάλληψη των αρκών ξηράς. Κυρία Υπουργή, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια εργάζεται για την πλήρη εξάλληψη των ε, ναρκών ε, ε, ξηράς κατά προσωπικού για να μπορέσει να λύσει τα ανθρωπιστικά προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Από το Μάιο του 1995 με την απόφαση που είχε λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την πρώτη κοινή ενέργεια για να καταπολεμήσει την χρήση και την ε, επέκταση των ναρκών ξηράς κατά προσωπικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ήταν η πρώτη ε, μέσα στην διεθνή κοινότητα που το 1997 ενήργησε μετά από την διάσκεψη της Ολτάβα και της συμφωνίας για την ε, μεταφορά των αρκών ξηράς κατά προσωπικού και στη συνέχεια η ε, Ευρώπη ανέλαβε μία νέα δράση για την πλήρη κατάργηση, πλήρη κατάργηση αυτών των αρκών ξηράς και για να υπάρξει ένα κοινό μορατόριο σχετικά με την παραγωγή αυτών των αρκών και την κάλυψη των πολλαπλών ενεργειών που χρειαζόταν για να μπορέσουν να αποδυναμωθούν οι μηχανισμοί αυτοί. Από το 2003 έχουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας και το 2008 αναλάβαμε ένα νέο κοινό μέτρο για να στηρίξουμε την παγκόσμια εφαρμογή ε, της συνθήκης της ΟΤΑΒΑ και να βοηθήσουμε συγκεκριμένα τα, κράτα, τα, τα κράτη που συμμετείχαν εις την συνθήκη αυτή ιδίως όσον αφορά αφορά την απομάκρυνση των αρκών και την καταστροφή των αποθεμάτων. Παρόλο που έχουν αυξηθεί τα κράτη που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία και μειώνεται το ποσοστό των αρκών ξηράς αυτών, ε, παραμένουν πολλά προβλήματα στην ζωή των θυμάτων και ε, στο πρόγραμμα 2010-2014 το οποίο υιοθετήθηκε στην Καρθαγένα της Κολομβίας στις 29 ε, Νοεμβρίου μέχρι 4 Δεκεμβρίου του 2009 το Συμβούλιο καταρτίζει ένα νέο πρόγραμμα δράσεως για να μπορέσει να συνδράμει τα θύματα ε, σε συνδυασμό με τις πολιτικές ενέργειες του Συμβουλίου και η βοήθεια της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της πολιτικής γυτνιάσεως μαζί με τις προσπάθειες των κρατών μελών οδήγησαν σε μία αύξηση της ε, βοηθείας Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τους στόχους αυτούς που έφτασε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το ίμιση της παγκοσμίου συμμετοχής. Ευχαριστώ. Κύριο Higgins. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα για την πλήρη απάστηση. Αναφέρθηκε στη σύμβαση της Οτάβας. Είχαμε και σύμβαση του Δουβλίνου όσον αφορά τις, τους, α, τους, τους διάφορους οπλισμούς διασποράς κλπ. 1,8 ε, δισεκατομμύρια ευρώ δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ευαισθητοποίηση για τι ε, νάρκε τη ΕΣΕΣ για την περίοδο μέχρι το 2007. Διέθεσε. Μόνο 1,5 δι τελικά δαπανήθηκαν από το ποσό που δόθηκε. Ποια είναι η πραγματικότητα, ότι οι χερσαίε νάρκε χρησιμοποιούν είναι βαρβαρικοί βάρβαρη πρακτική. Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν ή ε, ακροτηριάζονται το μήνα. Και θα πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να υπάρχει κάποια κίνηση και ευαισθητοποίηση σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος. Ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, δίκαιο έχετε. Δαπανίσαμε ένα δισεκατομμύριο, ενάμιση δισεκατομμύριο, δύο χιλιάδες άνθρωποι είναι ακόμα θύματα κάθε μήνα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί μόνη της να κάνει όλη τη δουλειά, κάνει τη μισή ήδη. Εξηγήσατε σαφώς πόσο έχουμε ευαισθητοποιηθεί όσον αφορά την ανθρωπιστική πτυχή, την ανθρώπινη πλευρά του προβλήματος. Δυστυχώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ πιο πολύ όσον αφορά τις λήψεις ε, αποφάσεων και όσον αφορά τον αφοπλισμό πιθανότατα εκεί μπορούν να γίνουν πολλά βήματα και κάνουμε προσπάθειες όσον αφορά αυτό το θέμα της απαγόρευσης ναρκοθέτησης με νάρκες κατά προσωπικού. Ευχαριστώ, ο Πρόεδρος. Έχω δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις. Κύριος Κέλλη και κύριος Ρούμπικ. Ο κύριος Ρούμπικ είναι πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Οι νάρκες ξηρά και στο μέλλον θα αποτελέσουν σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει ένα πρόγραμμα εκαθαρίσεως αυτών των ναρκών. Νομίζω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ε, οργανισμούς οι οποίοι ε, έχουν ερευνητικά προγράμματα για να επιλύσουν αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον συνάδελφό μου που έθεσε το ερώτημα και ευχαριστώ και το Συμβούλιο για τι πλήρε απαντήσει που μα έδωσε. Για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε ότι ήταν πολύ ενεργό η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει αυτή την ατυχή κατάσταση. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το Συμβούλιο, είναι ικανοποιημένο το Συμβούλιο όσον αφορά την αντιμετώπιση πλευρά Ηνωμένων Εθνών. Μήπω μπορούμε να συμβάλλουμε με καλύτερο τρόπο, μάλλον το ΟΗΕ να συμβάλλει με καλύτερο τρόπο, να κάνει κάτι παρόμοιο αυτό που κάνουμε. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο όποτε είναι έτοιμο, α δώσει την απάντηση, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου. Είναι συμπληρωματικά τα ερωτήματα. Θα απαντήσω το πρώτο ερώτημα βάσει της δεύτερης. Πράγματι, κάθε ερευνητικό πρόγραμμα για την αποναρκοθέτηση είναι κάτι ευπρόσδεκτο. Χρειάζεται στενή συνεργασία με τον ΟΗΕ και πάνω απ' όλα πρέπει να συμφωνήσουμε εντός του ΟΗΕ με εκείνους που αποτελούν αυτές τις αρχές. Είναι ένα έργο μακρόπνοο. Πρέπει να πιστούν άλλοι που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τα μέσα που πρέπει να επενδυθούν για την κατάρτιση τέτοιων ερευνητικών προγραμμάτων. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ας πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση της κυρίας Μπικεβιτσιούτε και αφορά τη δημιουργία κέντρου παρακολούθησης κρουσμάτων βίας κατά των γυναικών. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών είναι ένας κοινό στόχος για το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα δύο θεσμικά όργανα, όπως γνωρίζετε, εργάζονται για το θέμα αυτό εδώ και χρόνια και σε διάφορα πλαίσια. Υπενθυμίζω το ψήφισμα το οποίο εγκρίνατε πέρυσι Οπότε και γιορτάσαμε τη δέκατη επέτειο από το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών ε, που ε, θεώρησε ότι 25η Νοεμβρίου θα είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Σε αυτό το ψήφισμα καλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει πρόταση κοινοτικής πολιτικής ε, που θα είναι στοχευμένη και συνεκτικότερη ζητώντας από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό σύστημα για τη συλλογή δεδομένων. Όπως υπενθυμίζει η Ευρωβουλευτής, ε, τον προηγούμενο Μάρτιο το Συμβούλιο κάλεσε την Κομισιό να ε, συγκροτήσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Μία από τις προτεραιότητες που εντόπισε το Συμβούλιο σχετικά είναι η προετοιμασία για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου ε, για κρούσματα βίας κατά των γυναικών με βάση τις εφιστάμενες δομές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή εκπονεί μια νέα στρατηγική για τη βία κατά των γυναικών, η οποία θα αφορά επίσης τη δημιουργία αυτού του παρατηρητηρίου, αλλά προς το παρόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν γνωρίζουμε το ακριβές περιεχόμενο. Ελπίζουμε να λάβουμε τη στρατηγική αυτή εντός του επόμενου έτους, άρα είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε μια διαφορετική πρόταση ε, που θα χρειάζεται στη συνέχεια να υιοθετηθεί για τη δημιουργία αυτού του παρατηρητηρίου. Όπως καταλαβαίνετε το Συμβούλιο ως νομοθέτης μπορεί να παρέμβει μόνο όταν θα υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια τέτοια πρόταση θα εξεταστεί με το δέοντα τρόπο από το Συμβούλιο που θα συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο ως νομοθέτη για και όπως καταλαβαίνετε προς το παρόν είναι πρόωρο να προβούμε σε υποθέσεις ε, για τα σχετικά με το παρατηρητήριο παρακολούθηση κρουσμάτων βίας κατά των γυναικών ή και σε ό,τι αφορά την ε, έναρξη λειτουργίας αυτού του παρατηρητήριου. Κυρία Μπλινκεβιτσιούτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την απάντησή σας. Πάντως νομίζω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την ελπίδα ότι κάποια μέρα θα μπορούμε να συλλέγουμε δεδομένα για, την, ε, για τα κρούσματα βίας κατά των γυναικών. Θέλω μια διευκρίνηση κατά την άποψή σας. Με βάση τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή, αρκούν τα στοιχεία αυτά για να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Νομίζω ότι η προτεραιότητα αυτή δεν έχει επαρκώς ε, οριστεί ακόμη και γι' αυτό λοιπόν έχουμε και τόσα κρούσματα βίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντηση. Δεν είναι λάθος αυτό που λέτε. Σήμερα είναι δύσκολο να πούμε ότι για τη δημιουργία του παρατηρητηρίου αρκεί να βασιστούμε σε αυτά τα οποία έχουν ήδη μεμονωμένα τα κράτη-μέλη, έχουν ε, ως απογραφή από κρουσμάτων βίας, αναλογία, ποσοστά. Είναι μια αρχή βέβαια για να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά αυτό που περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια κατεύθυνση, μια μεθοδολογία, ένα σχέδιο για να μπορέσουμε να προβούμε σε μια εναρμόνιση σε επίπεδο 27 κρατών μελών ώστε να έχουμε ένα αξιόπιστο τρόπο απογραφής ε, των κρουσμάτων βίας, ε, της διάστασης που έχει το φαινόμενο, ώστε να μπορέσουμε στο, βαθμό του, στο μέτρο του δυνατού να χαράξουμε μία αποτελεσματική στρατηγική. Συμπληρωματική ερώτηση από τον κύριο Ρούμπικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και η κυρία Βόλης. Ε, έχουμε οργανισμούς ε, οι οποίοι ήδη ασχολούνται με το θέμα αυτό και σας υπενθυμίζω το γραφείο στη Βιέννη. Δεν θα ήταν δυνατόν να καλέσουμε εδώ την οργάνωση και να τη ζητήσουμε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και να προετοιμαστεί για να μην χρειαστεί να δημιουργηθεί ένα νέο όργανο και να αναθέσουμε στην οργάνωση αυτή στη Βιέννη την δραστηριότητα αυτή όπου υπάρχει έμπειρο προσωπικό και νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια καλή λύση. Α Ας απαντήσω. Όντως ευχαρίστως να χρησιμοποιήσω έναν ισχύοντα οργανισμό αντί να δημιουργήσουμε ένα νέο. Έχουμε ήδη αρκετούς οργανισμούς, δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε νέους. Και ελπίζω ότι στην εκπόνηση της τακτικής που θα μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περάσουμε από τις ισχύουσες δομές όπως παραδείγματος χάρη η οργάνωση της Βιέννης. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση του κυρίου Φερνάντες που αναφέρεται στα βιολογικά απόβλητα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι κατόπιν προτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκνινε ε, το ψήφισμα σχετικά με την πράσινη βίβλο της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων και ε, στις 6 Ιουνίου. Ε, εκεί η Επιτροπή έχει εκπονήσει μία ειδική πρόταση και μελέτη για τα βιολογικά απόβλητα και θα πρέπει να ολοκληρώσει μελέτης ως το τέλος του 2010. Θα μου πείτε ότι τελειώνει το 2010. Ζητάτε λοιπόν από την Επιτροπή να εξετάσει προληπτικά μέτρα τη δυνατότητα διαχωρισμού των ε, ε, αποβλήτων που μπορούν να αποδομηθούν βιολογικά κατά τρόπον ώστε να καθοριστούν οι προϋποθέσεις για τη σήμανση για την ε, ε, χώνευση των αποβλήτων αυτών. Το Συμβούλιο σημείωσε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ε, διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπεται να υιοθετηθούν τεχνικοί κανόνες για Ε, ε, των θεμάτων αυτών και να αναθεωρηθεί η απόφαση 86 του 2008 σχετικά ε, με τις βιολογικές ύλες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε το Σεπτέμβριο μία πρόταση κατά τρόπον ώστε να εξεταστεί το θέμα αυτό αφού ένα συνέδριο είχε διοργανωθεί και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο Συμβούλιο στις 14 Οκτωβρίου. Δηλαδή είναι πολύ φρέσκο το θέμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε μία οδηγία συγκεκριμένη που αφορούσε τα οργανικά απόβλητα για σαφήνεια και απλούστευση και για νομική ασφάλεια πιστεύω ότι αντί αυτή την νομοθεσία που μοιράζεται διάφορα κείμενα είναι καλύτερα να έχουμε μια ειδική οδηγία τι ούτω τρόπος μπορούμε να συμφωνήσουμε όσον αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μέχρι το 2020 για την ευφυή e e και βιώσιμη ανάπτυξη για την ανάπτυξη την ενταξιακή διότι έτσι θα έχουμε και περισσότερες θέσεις απασχόλησης, πράσινες. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος με προϊόντα υψηλή ποιότητα, θα μπορούμε να δημιουργήσουμε ε, λοιπάσματα υψηλή ποιότητα από αυτά τα απόβλητα και να έχουμε καλή προσέγγιση αφορά τη βιοπικιλότητα. Συμφωνεί το Συμβούλιο με μια ειδική οδηγία γι' αυτό και τι κάνει για να πετύχει αυτό το στόχο που ανέφερα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Ήμουν πολύ ήπια απέναντί σα, διότι έχουμε αρκετό χρονικό διάστημα στη διάθεσή μα, αλλά 30 δευτερόλεπτα υποτίθεται πρέπει να είναι η ερώτηση δευτερεύουσα. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο, λέει ο Πρόεδρο του Συμβουλίου για να μην επαναφέρεται στην τάξη στο τέλο τη παρέμβασή μου, αλλά το ερώτημα είναι αρκετά ενδιαφέρον, ενδιαφέρον θα έλεγα. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προτείνει, να μία προτείνει μια τέτοια ειδική οδηγία. Το Συμβούλιο κατανοεί ότι στην ανακοίνωση σχετικά με τα επόμενα στάδια τη διαχειρίσεω των βιοαποβλήτων τη Ενώσεω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαπίστωσε κενά όσον αφορά την παρούσα νομοθεσία κάτι που θα απαιτούσε ειδική νομοθεσία, αλλά ανακοίνωσε μια πρόταση τροποποίησης οδηγία που αφορά αυτά του χώρους ε, καθαρισμού, σταθμού καθαρισμού. Κατά τη διάρκεια τη εργασία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του 2009 διεφάνει ότι τα κράτη-μέλη είναι μοιρασμένα όσον αφορά την αναγκαιότητα ύπαρξη μια ειδική οδηγία που αφορά τα βιοαπόβλητα. Η απάντησή μου δεν θα είναι ναι ή ου. Εφόσον τα κράτη-μέλη είναι μοιρασμένα, το Συμβούλιο θα εξετάσει προφανώ με ενδιαφέροντο την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την οδηγία που αφορά τον καθαρισμό των αποβλήτων και κυρίω τα βιολογικά απόβλητα που προφανώς θα καλύπτονται από την εν λόγω πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Τα σχόλιά μου δεν απευθυνόταν σε εσά. Και τώρα περνάμε στην επόμενη ερώτηση ερώτηση της κυρίας Γκίνες για τον κίνδυνο διπλής ύφεση καθώς και τη σκοπιμότητα του στόχου περί 3%. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο βασικός στόχος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης παραμένει η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις συνθήκες θα πρέπει τα κράτη-μέλη να διεξάγουν μια συνεκτική εθνική πολιτική. Συνεκτική δηλαδή με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξη και με τις γενικές κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής. Το Συμβούλιο της 7 Σεπτεμβρίου συμφώνησε για την εισαγωγή από το 2011 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Βασικός στόχος αυτού του εγχειρήματο είναι το χρονοδιάγραμμα για την παρουσίαση του προγράμματος ε, στο, Σύμφωνο σταθερότητα και των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων να είναι τέτοιο ώστε να μπορέσει να υπάρχει η απαραίτητη δημοσιονομική πειθαρχία, μακροοικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη και συγχρόνως να διατηρηθούν οι μεμονωμένες διαδικασίες που είναι ξεχωριστές. Θα βελτιωθεί έτσι ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μπορέσει να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία και μακροοικονομική σταθερότητα. Με λόγω της ίδιας ακριβώς μέρημνας και σεβόμενη τις ε, αρχές ε, των συνθήκων, η Προεδρία προβλέπει κάποια μέτρα για να υπάρξει ανάκαμψη. Ταυτόχρονα όμως ε, χωρίς να πληγεί και η απαραίτητη δημοσιονομική, δημοσιονομική πειθαρχία. Η νέα στρατηγική Ευρώπη 2020 στρατηγική για την ευφυή ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με αλληλεγγύη στις 17 Ιουνίου εγκρίθηκε το Συμβούλιο αυτή στρατηγική, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις αυτές και προβλέπει τον επαναπροσδιορισμό των πολιτικών για την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα υπέρ της ανάπτυξης, υπέρ της απασχόλησης που θα εγγυώνται ταυτόχρονα και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Η στρατηγική Ευρώπη 2020, όπως γνωρίζετε, μεταξύ των μεγάλων στόχων περιλαμβάνει την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθήκων για την έρευνα, βελτίωση του ε, εκπαιδευτικού επίπεδου, όπως είπαμε και πριν, και τη κοινωνική ένταξη μεταξύ αυτών βέβαια και την καταπολέμηση της στόχης. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι ασυμβίβαστο αυτό με τους στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας και με τα μέτρα για την ε, βελτίωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η κυρία Μαγκίνες. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Περίμενα περισσότερες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ όμως. Το κόμμα του που είμαι μέλος, το Φίνα Γκέιλ, Γκέιλ υποστηρίζει το στόχο 3% όπως και τα σημαντικότερα κόμματα της, της Ιρλανδίας. Έχοντας στόχο και ημερομηνία την επίτευξη αυτών είναι ζωτική σημασία. Όχι μόνο για τα δικά μας συμφέροντα αλλά και για το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και προσέξτε το εξή. Μια έξοχη ομιλία που έγινε το πρωί από πρώην από τον Τζον Μπρούτον που ήταν φίλος του Κοινοβουλίου που μιλάει ειλικρινά για τις προκλήσεις αλλά και το τι μπορούμε να κάνουμε και τι μας περιμένει όσον αφορά αυτούς τους σκληρούς στόχους. Η Ιρλανδία έχει πολλά προσόντα που θα μα επιτρέψουν να πετύχουμε του στόχου, χωρί να υποφέρουμε. Θα υπάρξει πόνο, θα τα καταφέρουμε, θα χειριστούμε τον πόνο. Σχόλια θα ήθελα και ήθελα να υπογραμμίσω και να σα επιστήσω αυτή την ε, ομιλία, την προσοχή όσον αφορά αυτή την ομιλία. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, λέει πρόεδρο. αν έχει την καλοσύνη να απαντήσετε. Αναφερθήκατε στο Ιρλανδικό πρόβλημα. Κατανοώ. Είμαστε όλοι ευαίσθητοι. Κατανοούμε το Ιρλανδικό πρόβλημα η απάντηση που δίδω στο ερώτημά σας είναι μια απάντηση ευρύτατη όσον αφορά τα 27 κράτη-μέλη, διότι πρέπει να έχουμε συνεκτικές πολιτικές, πολιτικές νομισματικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, ε, πολιτικές ανάκαμψης και αλήθεια, κάποιοι προφανώς συναρτήσει της ε, χρέωσής τους, του ετήσιου χρέους, εδώ και δύο-τρία χρόνια, και από όταν εμφανίστηκε η κρίση θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες μεγαλύτερες από άλλους. Η Ιρλανδία περνά δύσκολες στιγμές πράγματι και πρέπει να το πιστέψετε ότι η Ευρώπη καταλαβαίνει τις δύσκολες στιγμές που περνάτε. Νομίζω ότι αρκετές χώρες τα περνάνε αυτά και τα περάσουν αύριο και η λιτότης δεν εμποδίζει την αλληλεγγύη και στο βαθμό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε επιτάπητος αυτή την εβδομάδα όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση πρόταση, βλέπουμε τη μέρημνα που υπάρχει να μην αφιεθούν στο περιθώριο κάποιες χώρες, μία από τις χώρες. Ξέρετε τι έκανε στην αλληλεγγύη, για, στα αλληλεγγύη η Ευρώπη στην περίπτωση της Ελλάδας, δεν συγκρίνουμε τις δύο χώρες, αλλά επουδενή η Ευρώπη δεν θα αφήσει εκτός διαδρομής ένα από τα 27 κράτη-μέλη, στην άκρη του δρόμου. Θα τα αφήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Αρκετοί έχουν ζητήσει να υποβάλουν συμπληρωματικέ ερωτήσει. Ξανά φοβάμαι ότι πρέπει να κάνω επιλογή και να λάβω υπόψη ποιο ήδη έχει πάρει το λόγο και να πετύχω και πολιτική ισορροπία. Συμπληρωματικέ ερωτήσει από τον κύριο Κράουλη και τον κύριο Παπα-Νικολάου. Ο κύριο Κράουλη είναι ο πρώτο που θα υποβάλει ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα για την απάντησή του. Δύο πράγματα θέλω να πω πολύ σύντομα. Καταρχά, όταν έγινε συζήτηση όσον αφορά το έλλειμμα του 3%, φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα λογιστικού υπολογισμού στα διάφορα κράτη-μέλη, σύμφωνα με κάποια κριτήρια. Δεύτερον, όσον αφορά την επιβολή των μέτρων, τι ευελιξία υπάρχει λόγω της παρούσης κρίσεως που πλήττει όλα τα κράτη-μέλη, περιθώριο για ποσοστό σφάλματος όσον αφορά το όριο του 3% που έχει τεθεί. Ο κ. Παπα-Νικόλα, έχετε το λόγο παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και στη στρατηγική για το 2020 βεβαίως υπάρχουν ε, μηνύματα τα οποία προσπαθούν να είναι αισιόδοξα. βεβαίω και στον προπολογισμό που ψηφίσαμε σήμερα σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων για το 2020 νομίζω ότι για παράδειγμα στην έρευνα και την καινοτομία δεν ανταποκρινόμαστε και δεν είναι δυνατό με αυτά τα μεγέθη να φτάσουμε στου στόχου που θέλουμε. Σιωπή όμω βλέπουμε από το Συμβούλιο σε σχέση με τι μεγάλε ανισότητε που υπάρχουν στο Βορρά και τον Νότο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω πρόσφατη δήλωση Κορυφαίου τελέχους και αξιωματούχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του προέδρου του eurogroup σύμφωνα με την οποία οι μεγάλε χώρε τη Ένωση, η γαλλία και η γερμανία ήξεραν το πρόβλημα τη Ελλάδο. το λέω αυτό επειδή αναφερθήκατε στην ελλάδα και παρόλα αυτά δεν έκαναν κάτι το προηγούμενο διάστημα γιατί είχαν μεγάλη ωφέλεια από την κατάσταση αυτή οι συγκεκριμένε χώρε. περιμένουμε κάτι κάποια πρωτοβουλία πιο συγκεκριμένη για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στο βορρά και τον νότο της Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις, δύο απαντήσεις. Σχετικά με την πρώτη ερώτηση. Βεβαίως, μέχρι τώρα, ακόμη και σήμερα, υπάρχουν ορισμένες διαφορές στα λογιστικά πρότυπα και η εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων προχωρά, διότι αν θέλουμε αύριο να μπορέσουμε να είμαστε ε, συνεπείς με τα κράτη-μέλη πρέπει να βασιζόμαστε στους ίδιους τρόπους υπολογισμού γι' αυτό και προχωράει η εναρμόνιση όσον αφορά η ευελιξία με το περιθώριο του 2-3% η ευελιξία ε, έχει ξεκινήσει από το 2009 την βλέπουμε το 2010 θα ισχύσει το 11 και το 12 κατά τρόπον ώστε τα κράτη να μπορέσουν να επανέλθουν σε μια υγιή δημοσιονομική πολιτική γιατί αν εφαρμόζαμε ε, επακριβώς και αυστηρά το 3% όλοι ε, φέτος θα ήμασταν εκτός του προτύπου της ε, δημοσιονομικής περιστολής. Οπότε χρειάστηκε τα κράτη-μέλη να έχουν χρόνο για να μπορέσουν να επανέλθουν σε αυτήν την δημοσιονομική αξιονομική ισορροπία μέχρι το 2013. Όσον αφορά την ανισότητα μεταξύ Βορρά και Νότου, είτε μιλάμε για ανισορροπία μεταξύ Βορρά και Νότου, είτε μεταξύ κρατών μελών που μάλλον βασίστηκαν στις ενισχύσεις που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναπτύξουν την οικονομία τους, να αναπτύξουν τον παραγωγικό ιστό, την απασχόληση και άλλοι που το έκαναν λιγότερο νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως υπάρχει για να διατηρήσει αυτή τη συνοχή και τα, ε, ε, ε, τα ταμεία τα οποία υπάρχουν στην Ευρώπη, ιδίω δε το Ταμείο Συνοχής που είναι το πρώτο κονδύλι στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αποβλέπει να μετριώσει αυτή την ανισορροπία μεταξύ, όπως είπατε, βορρά-νότου, αλλά δεν είναι η μόνη ανισορροπία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ ο κύριος Κούνατσεν σχετικά με την ερώτηση της κυρίας Τίκαου που θα είναι η τελευταία σήμερα σχετικά με την ελεύθερη διακίνηση, διακίνηση των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων και των εργαζομένων είναι ένα ουσιαστικό δικαίωμα και επιτρέπει εις τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ερώσεως να ζουν και να εργάζονται σε ένα άλλο κράτο μέρος. Εις τις συμφωνίες προσχωρήσεως προβλέπεται ότι τα κράτη πρέπει να αξιολογούν τις επιπτώσεις στην ε, εσωτερική αγορά και να μειώσουν τους περιορισμούς ή να τους καταργήσουν μέχρι στο τέλος της μεταβατικής περίοδου, δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο του 2011 για τις χώρες που προσχώρησαν το 2004 και 2013 για τις χώρες που προσχώρησαν το 2007. Ε, σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις προβλέπεται ότι θα αρθούν όλοι αυτοί οι περιορισμοί στην τρίτη φάση της μεταβατικής περίοδους διότι ε, διαφορετικά οι αγορές ε, ε, εργασίας θα υπέφεραν από σοβαρές ταραχές και γι' αυτό τα κράτη-μέλη ε, δεν έχουν προβεί σε αλλαγή του πλαισίου αυτού ενώ τα περισσότερα κράτη επιτρέπουν την ε, ελεύθερη προσχώρηση ε, στους υπηκόστων των χωρών που προσχώρησαν μετά το 2004 δεκα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ακόμη περιορισμούς και το Συμβούλιο είπε ότι η οικονομική κρίση δεν μπορεί να αναφέρεται για να επικαλείται κανείς την εφαρμογή αυτών των διατάξεων και καλεί τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν νέες δυνατότητες, να αναλύσουν τα εμπόδια εις την ε, ε, διακίνηση των εργαζομένων και να καταργήσουν τους, ε, τους υπάρχοντες περιορισμούς σύμφωνα με τις συνθήκες. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Τικάου τώρα και μία ε, επιπρόσθετη ερώτηση του κυρίου Παπα-Νικολάου, αλλά πρώτα η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα σας παρακαλέσω και εσάς και το Συμβούλιο να ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη να άρουν τους περιορισμούς και τους φραγμούς ε, στην ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων, ιδίως από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Να επισημάνω το εξής. Ίσες ευκαιρίες για την αγορά εργασία σε όλους τους εργαζομένους από όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης θα έχουν ως αποτέλεσμα την προστασία των εργαζομένων στις χώρες ε, προορισμού. Καλό λοιπόν τον Υπουργό να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να άρουν τους περιορισμούς που υπάρχουν στην ελευθερία. και πάλι το λόγο Κύριε Υπουργέ, από τη μία έχουμε τα προβλήματα σε ό,τι αφορά την κινητικότητα, από την άλλη έχουμε και τις πρωτοβουλίες της Ευρώπης για την ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζομένων που σε μια τόσο δύσκολη περίοδο είναι δεδομένο ότι αποτελεί μια επιλογή για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες, ιδιαίτερα του νέους ανθρώπους καταστρώσαμε το 2007 το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την κινητικότητα στην εργασία, το οποίο λήγει το 2010. Αναμένουμε μια αξιολόγηση για το σχέδιο αυτό και μια νέα πρόταση του Συμβουλίου. Έχουμε επίσης το πρόγραμμα Λεωνάρδο Νταβίνση για την ε, κινητικότητα των εργαζομένων. Αναμένουμε ενίσχυση αυτού του προγράμματος ή και νέες πρωτοβουλίες σχετικές. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια ακόμα συνάδελφος που θέλει να θέσει πληρωματική ερώτηση. Κυρία Σίνκλε. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα. Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κίνηση των εργαζομένων και συγκεκριμένα προσφύγων που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που παίρνουν χαρτιά για να μπορούν να μετακινούνται ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά και τη σύμβαση του 1951 για τους ετούντε άσυλο, τι βήματα, τι μέτρα έχει λάβει το Συμβούλιο σε σχέση με όλα αυτά. Πρόεδρος, μπορείτε να απαντήσετε κύριε Υπουργέ και τα τρία αυτά ερωτήματα μαζί. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι μια πραγματική προτεραιότητα του Συμβουλίου. Νομίζω ότι κάνουμε τα πάντα για να πούμε στα κράτη-μέλη που διατηρούν κάποιους περιορισμούς ότι πρέπει να αναλύσουν αυτή τη μεταβατική φάση στη διάρκεια τη οποία διατηρούν αυτού του περιορισμού και να δουν πώ μπορούν να τους άρουν, να άρουν αυτούς τους περιορισμούς. Πρέπει επίση να προσθέσω για να απαντήσω σε μία από τι ερωτήσει ότι αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι πράγματι πρωτοβουλία, ε, μάλλον προτεραιότητα του Συμβουλίου, αλλά συγκεκριμένα και τη Βελγικής Προεδρία. γιατί θα δείτε στο πρόγραμμα εργασία των 18 μηνών της ε, Τρόικας ε, των Προεδριών, Ισπανία, Βέλγιο, Ουγγαρία, ότι θα επεξεργαστούν όπως και επεξεργάζονται τις διατάξεις εσωτερικής αγοράς για την πραγματική εφαρμογή των τεσσάρων ελευθεριών, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό της εσωτερικής αγοράς. Στο πρόγραμμά μας λοιπόν εμείς συγκεκριμένα αναφέρουμε το ενδεχόμενο εξέταση ε, των των μετάβασης ε, για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που προέρχονται από τα νέα κράτη-μέλη. Τώρα, αυτοί οι μεταβατικοί περιορισμοί είναι ασυμβίβαστη με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Δεν ε, να σε μένα να προβώ σε αυτή την ε, αξιολόγηση. Οι περιορισμοί αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για όλες ε, τις Πέραν λοιπόν ε, τη παρότρινση που μπορούμε να εκφράσουμε για τα κράτη-μέλη ώστε να αναλύσουν τον αντίκτυπο που έχουν αυτοί οι περιορισμοί στην αγορά εργασία του ε, και να αποφασίσουν κατά πόσον θα άρουν αυτού του περιορισμού πριν τη λήξη τη μεταβατική περίοδου Απρίλιο 2011 και Δεκέμβριο 2013 για το 2004 και η ΔΕ για το 2006 δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο η Πρόεδρος. Ε, θα απαντηθούν γραπτώς οι υπόλοιπες ερωτήσεις και να σας ε, κάνω μια ανακοίνωση από την ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μου ζητήθηκε ο κύριος ε, Σαλόμ να συμπεριληφθεί στην Επιτροπή Σταγματικών Θεμάτων αντικαθιστώντας τον κύριο Ατόντο. Υπάρχουν σχόλια? Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν, επομένως εγκρίνεται ο διορισμός αυτός